προσβλέπω σε μια πιο δραστήρια και πιο συνεργατική προσέγγιση ε, μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Κυρία Μογκερίνη, επενέσατε την ευρωπαϊκή στρατηγική ε, ε, εσείς, επομένως επιτρέψτε μου να κάνω εγώ κάποιες επικρίσεις. Από ό,τι διαβάζουμε στην ιστοσελίδα τη Υπηρεσία εξωτερική δράση, αυτό θα αποτελεί ε, τρόπο για δράση σε δύσκολου καιρούς. Ε, αυτό το παραθέτω από την ιστοσελίδα. Έχω κάποια ερωτηματικά επ' αυτού. Πρόκειται για μια παγκόσμια στρατηγική χωρίς γεωγραφία. Πώς μπορείτε να έχετε παγκόσμια στρατηγική χωρί γεωγραφία. Δεν απαντά τελικά στην ερώτηση Ποιε πολιτικές είναι περισσότερο υποσχόμενε από άλλε και θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Υπ' αυτή την έννοια η στρατηγική δεν είναι καθόλου στρατηγική φύσεως. Επίσης, τονίζει την ανάγκη πρόληψης, ε, ε, επίλυσης και σταθεροποίησης. Αλλά όταν βλέπουμε τα προτινόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε κάτι εκ αντίθετο. Το πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο προτείνει περικοπή των περισσότερων δαπανών που είχαμε στο παρελθόν για αυτούς τους σκοπούς και είναι ένα απλό 40% των όσων είχαμε προηγουμένως. Πιστεύω λοιπόν, εάν πάρουμε στα σοβαρά τη στρατηγική, ότι θα πρέπει να ξοδεύουμε χρήματα για αυτά τα οποία υποτίθεται ότι πρεσβεύουμε. Και επίση ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε κατεπήγοντα θέματα για το κλίμα, τα οποία είναι εντελώ υποτιμημένα μέχρι τώρα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω στου αδέλφους να σεβαίνονται ε, σα παρακαλώ το χρόνο αγόρευση. Τώρα, εξ ονόματο ε, της ομάδας ID, Ταυτότητα και Δημοκρατία, ο κύριο Μαριανή για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία στο πλαίσιο της Ευρώπης των Εθνών, η οποία ε, δημιουργήθηκε ε, με βάση κυρίαρχα κράτη, ε, βλέπει μια πραγματική πολιτική και ανεξάρτητη πολιτική και θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το όρομα του στρατηγού Ντεγκόλ. Ε, σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ε, έλλειψη ισχύω ε, και πραγματικά έλλειψη ισχύω ενώπιον των Ισλαμιστικών κινδύνων, υποταγή στον, στα όσα υποτάσσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και δεν είμαστε ειρηνικοί, δρούμε όμως κατά των συμφερόντων των ευρωπαϊκών εθνών. Όσο τα τα πυρηνικά, δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη πολιτική ενώπιον της πολιτικής ε, στην, ε, ε, των ΗΠΑ, ενώ μόνο μία συνολική αποτελεσματική ε, πολιτική θα μας επιτρέπει. Ε, πού είναι οι ε, υποσχέσεις για την επανέναρξη των εμπορικών σχέσεων με το Ιράν. Λέτε, αυτή είναι η διάσημη ρητορική σας, ότι έχουμε πολιτική για τη Ρωσία και κάθε έξι μήνες ανανεώνουμε τα μέτρα για το εμπάργο χωρίς να εξετάζουμε το κόστος και τη δημιουργηματική του σημασία. Υπάρχουν καταστρεπτικές επιλογές για το πρόβλημα για τη Συρία. Ένας πρώην Υπουργό Εξωτερικών ε, εκφίασε και την καλή δουλειά που έκαναν ε, οι Αλκάιντα για τη Συρία και ε, ο γαλλικός στρατός είναι ο μόνος ο οποίος δίνει μάχη στην περιοχή του Σαχέλ. Και τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν καμία λύση στην πραγματικότητα. Δεν μπορείτε να δώσετε καμία φιλοδοξία για την Ευρώπη, γιατί το πρόγραμμα το οποίο διατηρείτε είναι απλώς ε, κάποιες τοπικές δράσεις ε, ε, που δεν λαμβάνουν υπόψη την νέα παγκόσμια τάξη. Ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ο λόγος στον κύριο Βάιμαρ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, ούτε ένα ε, κομμάτι της αξιολόγησης ε, που κάνατε για την παγκόσμια στρατηγική δεν αφιερώθηκε στον Ισλαμικό εξτρεμισμό ή την παγκόσμια δίωξη των χριστιανών. Αυτό πραγματικά είναι επέσχυντο Οι ριζοσπαστικοί μάμιδες ε, παίρνουν ε, εκατομμύρια ευρώ από, το κοινοτικό κορβανά και προωθούν ε, τη, τον διαχωρισμό των κοινοτήτων. Και παρόλα αυτά ενισχύουμε και βαθύνουμε τη συνεργασία μας με χώρες ε, που είναι πολύ επίκης και συγκαταβατικές απέναντι στον Ισλαμισμό. Και πολύ συχνά τέτοιε χώρες ανέχονται ή ενθαρρύνουν ακόμη τη δίωξη χριστιανών. Οι χριστιανοί περιθωριοποιούνται στην Μέση Ανατολή και εκδιώκονται. Και μάλιστα βλέπουμε σε μια μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου πώς ο εξτρεμιστικός Ισλαμισμός οδηγεί σε γενοκτονικέ δράσεις ει βάρο των χριστιανών. Οπότε η ε, αναπτυξιακή και εμπορική μας πολιτική θα πρέπει να σταματήσει την προώθηση του εξτρεμιστικού Ισλαμισμού και να προωθήσουμε, ε, να προστατεύσουμε ευάλωτες μειονότητες που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα της ΓΟΕ NGL, το λόγο έχει η κυρία Ζλέμ Ντεμιρέλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, αυτό που μας παρουσιάσατε ως παγκόσμια στρατηγική δεν είναι τίποτα άλλο ε. από μια, ένας κατάλογος ε, αυτά που θα θέλατε ε, για τη στρατιωτικοποίηση. Αυτά είναι κάτι που θέλει η Γερμανία και η Γαλλία και κάποιοι άλλοι. Εμείς ως αριστερά τα απορρίπτουμε. Θέλετε να αποκτήσει περισσότερες ε, στρατιωτικές δυνατότητε και να επιβάλλετε τη γεωστρατηγική σα πολιτική για τις εμπορικέ οδούς και για τους πόρους φυσικά. Και τα τελευταία χρόνια κάνατε πολλά πέσκο, στρατιωτική κινητικότητα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Είναι μόνο μερικά παραδείγματα από αυτά που διαπράξατε. Ε, δαπανίσατε δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς ενώ από την άλλη μεριά δεν έχουμε βρεφονιμπιακούς σταθμούς και 113 εκατομμύρια συμπολιτών μας ε, είναι στην παγίδα της φτώχειας. Εσείς θέλετε να δώσετε 30 δις τώρα για όπλα, για drone, drone δολοφόνους. Αν θέλετε να κάνετε κάτι για την ασφάλεια των συμπολιτών σας, να δαπανίσετε αυτά τα χρήματα για υποδομέ. Και επίση να κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποφύγετε ένα πόλεμο με το Ιράν και να ζητήσετε περισσότερε ε, συνθήκε αφοπλισμού. Αυτό θα ήταν στρατηγική υπέρ των λαών τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω, σα παρακαλώ, να σέβεστε το χρόνο σα. Και αλλιώ θα υποχρεώνομαι να σα κόψω το λόγο που είναι κάτι που πραγματικά δεν θέλω να κάνω. Και τώρα η κυρία, ο κύριος Νέιθον Τζιλ. Παρακαλώ. με μόνο εννέα ψήφους το Κοινοβούλιο σήμερα εξέλεξε με ένα ψηφοδέλτιο που είχε μόνο μία υποψήφια, την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Είναι μια υποψηφια την ουρσουλα φοντερ ειναι μια ευρωφανατικη που πήρε τη θέση της μέσω παζαριών και κλεισμένων των θυρών. Και όποια και, είναι, και όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντησή της είναι πάντα περισσότερη Ευρώπη. Και το λέει ανοιχτά. Θέλει να φτιάξει στρατό της Ένωσης και λέει ότι δεσμευόμεθα επίσης για τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Μα ένα από τα δύο. Δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήσουμε και τις δύο αυτές ε, προτεραιότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο ποτέ δεν πρέπει να καταλήψει την κυριαρχία του που συμπεριλαμβάνει τις ενόπλες δυνάμεις του. Ο Μπόρις Τζόνσον και η συντηρητικοί να είναι προειδοποιημένοι αν ε, παραδώσετε τις ένοπλες δυνάμεις μας σε έναν ενωσιακό στρατό της Ένωσης, ο λαϊκός στρατός του Βρετανικού Εκλογικού Σώματος θα σας τιμωρήσει στις κάλπες. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντούμπραφ Κασούιτσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Μακερίνη, χαίρομαι που η συζήτηση αυτή για την παγκόσμια στρατηγική μας είναι και η πρώτη συζήτηση που έχουμε στην νέα κοινοβουλευτική θητεία. Ε, είμαστε υπέρ αυτή τη στρατηγική που εδράζεται στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κράτο δικαίου και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Δυστυχώς δεν είναι ο κόσμος μας σε καλύτερη μοίρα από ότι το 2016 που ξεκινήσαμε τη στρατηγική, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις πολυμερείς πλατφόρμες για να προωθήσουμε την πολιτική μας ασφάλειας και άμυνας, εξασφαλίσουμε σταθερότητα και ειρήνη και να γίνει η παγκόσμια στρατηγική ε, η πηξίδα μας για την εξωτερική μας δράση στον κόσμο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να έχει από τα αποτελέσματα. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, περισσότερες και πιο στενέ εταιρικέ σχέσει. Όλοι περιμένουν από εμά ισχυρότερη Ευρώπη, κυρίω οι πολίτε. Αλλά όχι μόνο οι Ευρωπαίοι πολίτε, και ο υπόλοιπο κόσμο περιμένει ισχυρότερη Ευρώπη. Πολλέ φορέ τίθενται να ευρωπαϊκά σχέδια, ενώ εμεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ευημερία. Και αν δεν ξέρετε τον όρο τη δημοκρατία, θα ήθελα να πω στον προλαλήσατε, και μία ψήφο διαφορά σημαίνει δημοκρατία. Ευχαριστώ. Το λόγο η κυρία Σάντους για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν περάσει τρία χρόνια από την Παγκόσμια Στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχαίρω την κυρία Μαγκερίνη για την εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Ε, είμαστε υπέρμαχοι της πολυμέρειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το ισχυρό μας σημείο, αυτό είναι το ατού μας και θα ήθελα να ε, επισημάνω κάποια επιτάγματα της στρατηγικής, ε, τα προγράμματα στρατηγικής και ασφάλειας και ενισχυμένη μόνιμη συνεργασία, το ΠΕΣΚΟ, η συμφωνία για, την, για τις επενδύσεις στην Ουκρανία, η στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως και ένας τομέας όπου έχουμε να κάνουμε πολλά. Ο εσωτερικός και εξωτερικός άξονας των μεταναστευτικών ροών είχε κάποια αποτελέσματα με προγράμματα όπως το επιχείρηση Σοφία, αλλά δυστυχώς εκεί πολλά έχουμε να κάνουμε ακόμη. Ιστερούμε, θα πρέπει να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν ε, Πολλές χώρες αρνούνται να εφαρμόσουν τους ε, διεθνείς διατάξεις για το άσυλο και περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι πρώτων πυλών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τόσους ε, πρόσφυγες σε στρατόπεδα προσφύγων στη Λιβύη που υφίστανται, από απάνθρωπη μεταχείριση και βασανιστήρια. Πότε επιτέλους θα προωθήσουμε αυτή τη στρατηγική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που απαιτούμε σε άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κιούτσουκ για ένα λεπτό. Ο Ήλιαν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία εκπρόσωπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, σταθερή σας συμμετοχή και ε, ε, ενεργό συμμετοχή σας στη συζητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλά έχει πετύχει η παγκόσμια στρατηγική στην προάσπιση και προώθηση της πολυμέρης και της πολυμερούς παγκόσμιας τάξης και θέλουμε αυτό το στρατηγικό όραμα να το μετατρέψουμε σε απτή δράση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόοδο σε θέματα ασφάλεια και άμυνα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, βέβαια, γινόμαστε μάρτυρε πολλών συγκρούσεων σε πολλέ περιπτώσει και οι προσπάθειέ μα για την πρόθεση τη ειρήνη και τη ασφάλεια δεν στέφονται πάντα με επιτυχία. Από τη Συρία στη Λιβύη, τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Θα πρέπει να βρούμε τι σωστέ συμφωνίε για να καταλήξουμε σε βιώσιμε λύσει σε αυτέ τι πολύ σοβαρέ κρίσει. Επίση, θα πρέπει να θελοτυφλούμε απέναντι σε εκείνου ε, που εστερνίζονται τις αξίες μας και θέλουν να προσχωρήσουν στην οικογένειά μας. Η στρατηγική αναγνωρίζει την πρόοδο των Δυτικών Βαλκανίων, η Συμφωνία των Πρεσπών, η ε, μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη της Αλβανίας είναι σημαντικά θέματα, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να, αποκατασταθεί, για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή και να ενισχυθεί η ενταξιακή διαδικασία. Ευχαριστώ κύριο Σμπέρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρο, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύρια Μογκερίνη, η τέχνη του πολέμου, λέει ο Σούντσου, είναι ότι πρέπει τα σχέδιά σου να τα εκπονείς σε, απόλυτη αδιαφάνεια τη νύχτα και μετά να δράς ως αστραπή. Το πρώτο το καταφέρνετε, αλλά το δεύτερο δεν το καταφέρνετε. Το κείμενό σας έχει πολλούς φιλόδοξους στόχους, αλλά δεν είναι το περιεχόμενο που με ανησυχεί είναι το θέμα της εφαρμογής. Από τότε που υπάρχει αυτή η παγκόσμια στρατηγική, ο κόσμος είναι χειρότερος. Μας βοηθάει λοιπόν η στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις κριτικές προκλήσει. κρίσιμες προκλήσεις. Η εξωτερική πολιτική ε, μας φέρνει σε σύγκρουση με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Στις προηγούμενες ευρωεκλογέ ήταν σαφές ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος ανησυχεί για την διάσταση της μετανάστευση. Όμως η στρατηγική σας οξύνει περαιτέρω αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό να έχουμε μια στρατηγική ταχεία αντίδραση που να βασίζεται στα συμφέροντα των κρατών μελών. Να εργαστούμε προ αυτή την κατεύθυνση, ούτω ώστε οι σχέσει μα με σημαντικού άλλου παράγοντε όπω η Ρωσία και οι ΗΠΑ να βελτιωθούν. Πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική πολιτική για τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Μακάλιστερ, ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατήκ, εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Τρεις, ε, τρία χρόνια μετά τις πέντε προτεραιότητες ε, του 2016 για την παγκόσμια στρατηγική εξακολουθούν να παραμείνουν ε, ισχυρές αυτές οι, προτε, ε, προτεραιότητες. Προσέγγιση για τις συγκρούσεις, ε, συνεργατικές περιφερειακές ε, προτάσεις και αποτελεσματική κυβέρνηση. Εγώ είμαι υπέρ της αυξημένη ε, συνεργασίας για την άμυνα μεταξύ των κρατών μελών και τα βήματα τα οποία λήφθησαν για να έχουμε στρατηγική αυτονομία. Η συνολική εφαρμογή βέβαια της στρατηγικής έχει περιθώρια βελτίωσης χωρίς καμία αμφιβολία η ε, πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνδυάσει καλύτερα πολιτική σε εργαλεία που αφορούν τη διπλωματία, την ασφάλεια, την άμυνα, ε, χρηματοδότηση, ανάπτυξη του εμπορίου κλπ. Και επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε και την ευελιξία των εξωτερικών μέσων χρηματοδότησης και τέλος ε, θα πρέπει να έχουμε και πλειοψηφία και συγκεκριμένου τομεί τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Χαίρομαι που η νέα πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ούρσουλα von το ανέφερε σήμερα το πρωί στην παρέμβασή τη και να ευχαριστήσω την Φοντερίτα Μογκερίνη για την πολύ καλή δουλειά που έκανε σε αυτή την παγκόσμια στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Μπενιφέη για ένα λεπτό. Μπράντο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με, ενώ εσείς κυρία είπατε εκπρόσωποι εργάζεστε σε ένα διεθνές πλαίσιο μεγάλης αβεβαιότητας αναδύονται κάποια ανησυχητικά στοιχεία για την ε, ε, κίνηση κάποιων ε, ανθρώπων που βρίσκονται πάρα πολύ καλά στη λίγα του Ματέο Σαλβάνδίνη για να συσφίξουν σχέσεις με ε, σκοτεινούς πόρους χρηματοδότησης από την Ρωσία. Αυτό αποτελεί το σημαντικό πλαίσιο μιας εξωτερικής πολιτικής που αφορά την κοινή ευρωπαϊκά άμυνα, την στρατηγική αυτονομία, ακόμα και ε, ε, με βάση το ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι τώρα αν θα συνεχίσουμε αυτή την αυτονομία ή θα υποκύψουμε σε συγκεκριμένες δυνάμεις. Όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία ανέκυψαν στην Ιταλία και όχι μόνον, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν τα όσα έκανε η Task Force Stratcom και να συστήσουμε μια ερευνητική επιτροπή για το τι κάνουν η ακροδεξιά με την ε, Μόσχα ε, για και καλυμμένες πολιτικές κινήσεις. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή που αναδύεται ως πραγματικότητα πραγματική απειλή και το τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος ε, στον κύριο Γκετά για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπέτη εκπρόσωπε, παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες ε, που σας ε, περιποιούν τιμή και παρά τα πολλά επιτέγματα για τα οποία σας συγχαίρω, η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία η ευρωπαϊκή δημοκλα... διπλωματία πασχίζει να ακολουθήσει τις εθνικές διπλωματίες ε, σε ό,τι αφορά τη βαρύτητά της στο διεθνές προσκήνιο. Και αυτό δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί ε, φαίνεται ότι προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις για μια κοινή άμυνα, κάτι που προϋποθέτει κοινό όραμα για τα συμφέροντά μας, ε, τη θέση μας στον κόσμο και τις απειλές και κινδύνους που καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε. Πού βρισκόμαστε σε όλες αυτές τις συνθήκες η θα μπορούσε να έχει ως βασική αποστολή και βασικό καθήκον να προσδιορίσει καταρχήν τους μέσο και μάκρο μακροπρόθεσμους στόχους μιας ευρωπαϊκής διπλωματίας, δεύτερον τα μέσα ε, μιας τέτοιας σύγκλησης και τρίτον τα στάδια που θα προϋπόθεται κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ και περιμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μιγιάν Μον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η στρατηγική ασφάλειας ε, κατέδειξε τη σημασία μιας ε, ενεργούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε εξωτερικές σχέσεις. Η απομόνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνεται καν στις επιλογές μας σε έναν πολυμερή και διασυνδεδεμένο κόσμο. Αλλιώ απομονωμένοι θα ήμασταν αδύναμοι και εν τη ενώση ισχύς σίγουρα. Η εξωτερική μας πολιτική χρειάζεται, όπως είπατε και εσείς κυρία είπατε εκπρόσωπε, πολιτική βούληση. Προϋποθέτει πολιτική βούληση, δηλαδή ακράδαντη πεποίθηση ότι θα δράσουμε καλύτερα να δράσουμε από κοινού. Σήμερα όμω έχουμε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό και ελοχεύει ο διχασμό. Και η λήψη αποφάσεων επίση επιβραδύνεται. Και γι' αυτό, σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και το, τα εμπόδια που δημιουργεί η διαδικασία της ομοφωνίας. Βέβαια, θετική είδηση των τελευταίων χρόνων είναι τα επιτεύγματα στην πολιτική άμυνα. Κάτι που ζητούσαμε εδώ και χρόνια. Έχουμε περίπλοκο κόσμο, συγκρούσει, σειράξει, εντάσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μία μόνο ήπια δύναμη. Ε, φυσικά θα πρέπει να διατηρήσουμε τους, τους δεσμούς μας με το ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε ταυτόχρονα και τη δική μας αμυντική διάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Κάλιουραντ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και για την προσπάθειά σας. Όμως, ε, ένας από τους βασικούς τομείς της ε, στρατηγικής μας είναι η κυβερνοασφάλεια. Οι προκλήσεις στον χώρο αυτό είναι νέα πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τους κυβερνοκινδύνους και τις κύβερνο-απειλές διατηρώντας μια, ε, τον κυβερνοχώρο ανοιχτό, ελεύθερο και ασφαλή. Αναφέρατε διάφορα σημαντικά βήματα, τη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, την, ε, το, την εργαλειοθήκη για την ε, κυβερνοδιπλωματία, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και τονίζω τα εξή σημεία. Πρώτον, η Ένωση πρέπει να είναι παγκόσμια πιο ενεργή και να είναι πρωτοπορία και η κύρια φωνή στις συζητήσεις για την κυβερνοασφάλεια και τις δράσεις. Δεύτερον, η Ένωση πρέπει να πει περισσότερα, να γίνεται πιο ακουστή η φωνή της για έναν κυβερνοχώρο που να βασίζεται σε ρόλους. Ιδιαίτερα πρέπει να εφαρμόζεται ο διεθνής ε, νόμος και στο κυβερνοχώρο και πρέπει να πούμε περισσότερα για να μην εξαιρείται κανένας. Να ακούμε σε όλους και συνεργαζόμεθα με όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, Πάιτ, παρακαλώ, ένα λεπτό. Αγαπητή Φεντερίκα Μογκερίνη, έχουμε διάφορα θέματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στον κόσμο. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί το Συμβούλιο Ασφαλής των Μένων Εθνών, να αντιμετωπίσουμε την ε, κλιματική αλλαγή, συμφωνίες ελέγχου των, ε, ε του, εμπορί, εμπορίου όπλων. Πολλοί τομεί πρέπει να σε απασχολήσουν για να μπορέσει η Ένωση να είναι αποτελεσματική στο ρόλο της. Η ενίσχυση της κοινή πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας όλα έχουν γίνει από τότε που το συζητήσαμε στην Παγκόσμια Στρατηγική πριν από μερικά χρόνια. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα η ΠΕΣΚΟ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα και άλλα. Αυτό ε, αφορά και τον κυβερνοχώρο, την κυβερνοασφάλεια. Δυστυχώ η κλιματική αλλαγή θίγει και περιοχές που μέχρι στιγμής ήταν ήρεμες όπως η Αρκτική. Πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο και να αναπτύξουμε τη στρατηγική μας ούτως ώστε οι εντάσεις στην Αρκτική να μην αυξηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ζέλια Ναζόφκο για ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη είπατε εκπρόσωπε, χαίρομαι για την έκθεση εφαρμογής ε, της ε, παγκόσμιας ε, στρατηγικής και την ανάγκη που τονίζεται για συνοχή μεταξύ των πολιτικών μας και την ανάλυση των επιτευγμάτων μας. Θα πρέπει πολλά να πεδίσουμε ακόμη και παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, περισσότερο από ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια φιλόδοξη εφαρμογή της στρατηγικής για να ανταποκριθεί στις αλλαγές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσουμε μια παγκόσμια τάξη που θα εδράζεται στη δικαιοσύνη. θα πρέπει να έχουμε κοινέ αξίε και συμφέροντα για να υιοθετήσουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην πολυμέρεια. Καλωσορίζω ιδιαίτερα στη δράση μου για τη βελτίωση των σχέσεών μα με του ε, γειτόνου μα προ Ανατολά και προ τον Νότο. Να επικεντρωθούμε στη συνεργασία με τι περιοχέ αυτέ και κυρίω με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η, ειρήνη και η σταθερότητα εκεί δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένε. Θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα βήματα προ την διεύρυνση ε, και την ενταξιακή προοπτική αυτών των χωρών, γιατί θα είναι σημαντικά για την Ευρώπη στο σύνολό τη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πίτσουλα για μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε έχουν γίνει από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα Τα τελευταίων τριών ετών όμω είναι η οικοδόμηση τη Ευρωπαϊκή Άμυνα και κυρίω το οφείλουμε σε εσά. Θέλω να σα ευχαριστήσω για τη σημαντική δουλειά. Να έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα σε λίγα χρόνια παρά σε δεκαετίε και φαίνεται ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να κάνουμε πολλά. Έχουμε κάνει μια σειρά βημάτων προ να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Άμυνα πιο αποτελεσματική αφορά, την ευγνωστοποίηση των πόρων, να προστατεύσουμε του πολίτε μα καλύτερα, ενώ θα ενισχύσουμε τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω. Επίση, είναι σημαντική συμφωνία η πυρηνική με το Ιράν και εδώ πρέπει να βάλουμε τη δυνατά μα να τη διατηρήσουμε. Θέλω να αναφέρω ε, και τη συμφωνία των Πρεσπών, σημαντικό επιτεύγμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ελπίζω να την τιμήσει το Συμβούλιο και να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία φέτος ήδη. Όταν σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε τη σημασία της πολυμερούς τάξης. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να διατηρήσουμε τα προηγούμενα επιτεύγματα και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για το μέλλον. Η καλή τάση θα πρέπει να συνεχιστεί και να υποστηριχθεί με τους κατάλληλους πόρους που θα κατανοηθούν για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να δραματίζει ρόλο γιατί είναι σημαντική η soft power, θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία με τους συμμάχους μας και βοηθά στο να διατηρήσει και να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ειρήνη σε πολλά μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο ο κύριος Αλεξάνδρο Βιόρντανοφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μογκερίνη, η ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να συνιστά απειλή όχι μόνο για την ασφάλεια της ε, Βουλγαρίας αλλά για όλη την, την ασφάλεια όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατοχή στην Ουκρανία ήταν ευκαιρία για περαιτέρω επιθέσεις. Ο υβριδικός πόλεμος της ε, Ρωσίας εξαπολύεται και κατά της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικά, ε, σημαντικό για την ασφάλεια της Ένωσης να ενισχυθούν οι παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης, να ενισχύσουμε τα δυτικά Βαλκάνια και να επιταχύνουμε τις δραστηριότητες για την ενσωματωξή τους. Ελπίζω ότι θα ενταχθούν σύντομα στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τη Σερβία ιδιαίτερως. Η πολιτική της διεύρυνσης έχει μεγάλη δύναμη. και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ε, σύνδεσμο μεταξύ, στο συσχετισμό μεταξύ της συμμετοχής ενός κράτους στο ΝΑΤΟ και την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στη διαδικασία Catch the έχοντας ολοκληρώσει τις ε, παρεμβάσεις. Έχω τέσσερα αιτήματα με την κυρία Νίνα Τζιλ πρώτα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είπατε οι εκπρόσωπε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να δώσω έμφαση σε ένα σημείο της τελευταίας έκθεσης προόδου μεγαλύτερη ένωση, η ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά έχει μεγάλη σημασία. Θέλουμε να είμαστε σε ισότιμη βάση και να διαπραγματευόμαστε, να διαπραγματεύονται οι ηγέτες μας ισότιμα με τους άλλους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε όσο καλά και αν όλα αυτά που μας είπατε. Πρέπει να προστατεύσουμε την ε, πολυμερή συνεργασία ε, και βέβαια απαραίτητο αυτό θα είναι και ε, να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση του συστήματος των διεθνών οργανισμών. Η ασφάλεια βεβαίως έχει κέρια σημασία σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξει και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να στραφεί πλέον και να εξετάσει τον κίνδυνο που συνιστά η Κίνα όλο και πιο επιθετική στην Αφρική, τον Ειρηνικό αλλά και σε, άλλους, σε άλλες περιοχές του κόσμου καθώς οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνονται να οπισθοχωρούν από την πολυμερή συνεργασία και πρέπει να ανοίξουμε να τίνουμε και χείρα βοηθεία και να ανοίξουμε επιστολέ διαπραγματεύσει με την Αυστραλία, τον Καναδά και άλλε χώρε που συμμερίζονται τι αξίε μα και επειδή τελείωσε ο χρόνο μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να σέβεστε αυστηρά το χρόνο γιατί στο κάτω δεν θα προλάβω να δώσω το λόγο σε άλλον. παρακαλώ. Uh, we Εμεί, οι φιλελεύθεροι δημοκράτε από το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, το πιο σημαντικό ε, οικοδόμημα ειρήνης ε, στην ιστορία μας, αλλά πέραν της Ευρωπαϊκή ειρήνης θέλουμε μια παγκόσμια διεθνή τάξη συνεργασία, εμπιστοσύνη και συνεργασία ε, παγκοσμίω. Και αυτό το οικοδόμημα πλέον τίθεται να αμφιβόλο και εξαιτία τη μιλιταριστική τάση τη Κίνα και εξαιτία των ενεργειών τη Ρωσία του κυρίου Πούτιν, αλλά όλο ένα και περισσότερο ευθύνεται και η μη αξιόπιστη στάση των ΗΠΑ. Και αυτό κατέστη ιδιαίτερα σαφές από ε, τις ενέργειες του Προέδρου Τραμπ για το Ιράν. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που είχαν υπογράψει και οι ΗΠΑ και άλλοι σημαντικοί φορείς. Ο Ντόναλτ Τραμπ ουσιαστικά προωθεί την διάδοση των πυρηνικών όπλων με αυτή του την ε, προσέγγιση και είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου ε, και της συμφιλίωσης και υπεράσπισης αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Υπάρχει μία μπλε κάρτα από τις συναδελφορών, δεν Δέχεστε, κύριε Χόργουντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Είστε διατεθειμένος να ε, διακινδυνεύσετε τις ε, δομές που μας έχει δώσει τα τελευταία 70 χρόνια το ΝΑΤΟ για να διασφαλίσετε την ειρήνη ε, σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Γιατί θα, θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία να διακινδυνεύσετε πιο σημαντική διατλαντική σχέση απάντηση. Κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα όχι η κυρία Μογκερίνη δεν έχει αμφισβητήσει τη σημασία και αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ. Ακριβώ επειδή θέλουμε μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση στι απειλέ που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον κίνδυνο, όλα ε, και πιο επικίνδυνο κόσμο, γι' αυτό και χρειαζόμαστε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Ποιο αμφισβητεί το ΝΑΤΟ, ο πρόεδρο Τραμπ. Ε, που περισσότερο πρόσχεται στη, στη δική σας ιδεολογία ε, και το δικό σας λεκισμό από οποιοδήποτε άλλον. Ευχαριστώ. Λόπες Αγγιλάρ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, μόλις σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την κυρία Φόντερ Λάιεν ως νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι η δική σας θητεία θα ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι και να μένετε να αντικατασταθείτε από έναν έμπειρο ε, Υπουργό Εξωτερικών, τον Ζωζέ Μπορέλ, όπω ήσασταν και εσεί. Όμω θέλω να σα χαιρετήσω για τι προσπαθίε σα, για τα αποτελέσματά σας ε, και για την αφοσίωσή σα. γιατί ε, οικοδομήσατε αυτή την παγκόσμια στρατηγική στην Ισπανία. Όταν λέμε στρατηγική δεν την εξηγούμε, την εφαρμόζουμε και αν υπάρχει ένα τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει μια παγκόσμια στρατηγική, αυτή είναι η Αφρική. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημογραφία και το μεταναστευτικό. Χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια καθολική στάση απέναντι στην Αφρική. Και αν αυτό σημαίνει ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Και αν δεν είχε νόημα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Αφρική, θα πρέπει να το πράξουμε αυτό και να έχει ένα ρόλο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γουέρτ, παρακαλώ. Πρόεδρε. Θέλω να διορθώσω κάτι σε ό,τι αφορά ε, τις βλακίες που λένε ε, οι εθνικιστές. Ε, καταρχήν ε, έχουμε το Σουηδό βουλευτή Βένας, ο οποίος έδειξε άγνοια. Το 2017 συνάντησα Βρετανούς διπλωμάτες στην Κένια που με ενημέρωσαν για βασική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτρέπει τους εξτρεμιστές της να διασχίσουν τα σύνορα με τη Σομαλία και τους εμποδίζουν να έρθουν στην Ευρώπη και χαίρομαι που συλλογικά εμείς εκπαιδεύουμε αυτή την τοπική συνοροφυλακή. Η Βρετανοί εξωματούχοι μου ήταν αυτό, έτρεμαν μπροστά στην προοπτική του Brexit, καθώς υποσκάπτει την παγκοσμία και την εθνική ασφάλεια. Δεύτερον, ο Νέιθαν Γκέιλ, που είναι υπέρ του Brexit, ε, ε, παρουσιάζεται ως ε, πατριώτης πρωταθλητής για τις ενόπλες δυνάμεις της Βρετανίας. Όμως ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η εμπειρία ε, τους ε, να υπηρετούν σε όλο τον κόσμο και να συνεργάζονται με τους Ευρωπαίους εταίρους ε, τους εμπόδισε ε, να μη συμμετέχουν στην εκστρατεία για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παγκοσμία ειρήνη και ασφάλεια. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία 18 χρόνια το καθεστώς των ΗΠΑ και η Δυτική ε, συμμαχοί του κατάφεραν σημαντικά πλήγματα καταστροφικά σε όλο τον κόσμο, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη, την Ιεμένη. Τίποτε δεν δικαιολογεί τις πράξεις αυτές. Η Ευρώπη δυστυχώς έμεινε σιωπηλή δίστασε να τους καταδικάσει πολέμους για τους οποίους δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και τώρα βλέπουμε μια ε, ενίσχυση της έντασης ε, και της επιθετικότητας κατά του Ιράν, ένα είδος ε, πολεμικών επιχειρήσεων και μάλιστα το χειρότερο βλέπουμε να αναπτύσσεται εις βάρος του Ιράν και διερωτώ με η Ευρώπη τι κάνει. Θέλετε οι Σαουδάραβες και το Ισραήλ να εξαναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξουν σε πόλεμο με το Ιράν. Δεν μπορείτε να ε, ε, βοηθήσετε ώστε να ξαναγυρίσει η εθνική κοινότητα του Ιράν. Τι είναι αυτά με τις κυρώσεις. του Ιράν θέλει ειρήνη και όχι πόλεμο. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται έτσι τη διαδικασία Καρστιάη. Και δίνω το λόγο στην έπατη εκπρόσωπο, κυρία Μογκερίνη, για την απάντηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι εκτίμησαν και την παγκόσμια στρατηγική που παρουσίασαν πριν από τρία χρόνια και με τη στήριξη του Κοινοβουλίου πριν από τρία χρόνια, αλλά και την όλη δουλειά που κάναμε με το προηγούμενο Κοινοβούλιο για την υλοποίησή της. Σας ευχαριστώ που αναδείξατε την ανάγκη αφενός ε, να συνεχίσουμε ε, αυτή τη δουλειά, αλλά και να είμαστε συνεπείς ως προς αυτήν. Ας ξεκινήσω από το πιο άμεσο καθήκον για όποιον θέλει να είναι συνεπής ως προς την ανάγκη ε, να παραμείνουμε ένας ε, ε, αξιόπιστος παγκόσμιος παίκτη ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που προαναφέρθηκε που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι πρέπει ακριβώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε διακηρύξει. Να σα αναφέρω ορισμένα στοιχεία. Ω προ το ΠΔΠ συγκεκριμένα, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να αυξήσουμε του πόρου για την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατά 30% περίπου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο σε μια περίοδο αβεβαιότητα ανά τον κόσμο. Γιατί οι υπόλοιποι στρέφονται προς την Ευρώπη ε, στην προσπάθεια εξέβρεσης ενός αξιόπιστου, συνεργάσιμου ε, συνεταίρου κάποιου που πάντα επενδύει στη δημοκρατία και τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Όμω για να γίνει αυτό και να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια απαιτούνται και οι κατάλληλοι πόροι. Ελπίζω λοιπόν ότι και εσείς θα εργαστείτε προς αυτήν την κατεύθυνση τους επόμενους μήνες, ιδίως ό,τι αφορά την πρόταση που έχουμε κάνει με αύξηση κατά 23% για τους πόρους για την Αφρική. Πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας με την Αφρική ε, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και την πολιτική συνεργασία και εταιρική σχέση για την ειρήνη και την ασφάλεια, που πρέπει να τεθεί ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο του έργου μας στο μέλλον. 25% αυτών των πόρων αφορούν την κλιματική αλλαγή στην πρότασή μας. Ελπίζω και αυτή η πρόταση να τύχει τη στήριξή σας ε, κατά τις συζητήσεις για το επόμενο ΠΔΛΤΑΠΗ. Δεν θέλω να σχολιάσω την κατάσταση για το Ιράν, γιατί θα κάνουμε στη συνέχεια συζήτηση ακριβώς για αυτό το θέμα. Για όσους βέβαια θέλουν να παραμείνουν απόψε στο ημικύκλιο, σε ό,τι αφορά λοιπόν την κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Να τονίσω κάτι που γνωρίζετε ήδη, ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ελογικά να διατηρήσουμε την ε, συμφωνία με το Ιράν και να αποφύγουμε τυχόν κλιμάκωση και αντιθέτως να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό το διακύβημα από πλευράς ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κλιματική αλλαγή και διπλωματία. Να πω ότι και ένας άλλος τομέας, μάλλον, ε, προτεραιότητας για μας είναι η κυβερνοασφάλεια. Η ασφάλεια εν γέννη, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά και πιο συγκεκριμένα Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις στη στρατηγική και την έκθεση της στρατηγικής που θεωρώ ότι μπορούν να προωθηθούν επιτυχώς στο μέλλον. Δύο πράγματα ακόμα. Πρώτον, κάποιοι είπαν ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνση. Η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια αξιόπιστη διεύρυνση, πολιτική διεύρυνση και προοπτική διεύρυνση για τα Βαλκάνια. Αν και ο όρος διεύρυνση για εμένα δεν είναι σωστός, γιατί όλες αυτές οι χώρες είναι γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει λοιπόν με τη συμφιλίωση και ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, περιοχή. Ιδίω σε ό,τι αφορά την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Έχει έρθει η ώρα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να ληφθεί η απαραίτητη απόφαση από το Συμβούλιο του επόμενου μήνε το αργότερο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την δική μας ε, ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία. Να πω επίσης ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση ε, σε ό,τι αφορά τον χώρο τη μετανάστευση είναι κάτι που έχουμε συζητήσει αρκετέ φορέ εδώ στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου τους περασμένους μήνες, στην προηγούμενη θητεία. Μιλήσατε για το καλό έργο της επιχείρησης Σοφία. Νομίζω ότι γενικά έχουμε κάνει καλή δουλειά. Θυμάμαι όταν έφτασα εδώ πριν από πέντε χρόνια, η μετανάστευση δεν αποτελούσε αντικείμενο εξωτερικής πολιτικής, ήταν μόνο ε, κομμάτι της εσωτερικής μας πολιτικής. Νομίζω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε διαμορφώσει καλές σχέσεις ε, ε, με τους εταίρους μας. Έχουμε καλή συνεργασία και με τους οργανισμούς του ΟΗΕ, ιδίως την Υπατιαρμοστία για τους πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Και έχουμε και μία βιώσιμη προσέγγιση με τους εταίρους μας στα εξωτερικά μας σύνορα. Από την άλλη πλευρά, αν ε, κάτι με λυπεί είναι ότι η επιχείρηση Σοφία που κατάφερε να έχει ε, να καταπολεμήσει τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο τους ε, διακινητές, να κατάσχει σκάφη διακινητών, να σώζει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη αποφάσισε να απομακρύνει τα στοιχεία του ναυτικού, τα σκάφη στη Μεσόγειο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το αρνητικό. Πρέπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αποκαταστήσουμε την κατάσταση σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή και για την κατάσταση στη Λιβύη αλλά και για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τα δίκτυα διακινητών σε όλη τη Μεσόγειο. Τέλος. Ε, ακούσαμε κάποια, κάποιους προβληματισμούς και επικρίσεις για τον κίνδυνο στρατιωτικοποίησης ε, της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Ο δρόμος προς την ασφάλεια ποτέ δεν είναι επιθετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπαν κάποιοι από εσά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ένα, το, πιο επιτυχημένο μάλλον ε, project ειρήνη στην ανθρώπινη ιστορία. Καταφέραμε να επιλύσουμε τι εσωτερικέ μα ε, κρίσει και προβλήματα και με βάση αυτή την εμπειρία προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε τους εταίρους μας στη δική τους προσπάθεια ανέβρεσης λύσεων. Αυτό ισχύει και για ε, τις στρατηγικές μας δυνάμεις, αλλά και για τις ε, αστυνομικές δυνάμεις που συμμετέχουν ε, στις αποστολές μας. Τι κάνουμε ουσιαστικά, υποστηρίζουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς των χωρών εταίρων για να οικοδομήσουν θεσμούς ε, που θα ενισχύουν την ε, ασφάλεια, την άμυνα, είτε από πλευρά στρατιωτικών δυνάμεων, είτε σε πολιτικό επίπεδο για την θέσπιση, εγκαθίδρυση της ειρήνης, την λειτουργία των θεσμών στο επίπεδο της ασφάλειας και άμυνας υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ επισκέφθηκα τον Ήγυρα, την ε, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το Μαλί, αλλά αν δεν ήταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εκεί, αυτές οι χώρες ε, ε, θα αντιμετώπιζαν πολύ δυσχερέστερες συνθήκες. Επομένως, το δικό μας έργο δεν είναι ποτέ να σκοτώσουμε, ποτέ να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο καμία σύγκρουση. Αντιθέτως, ο δικός μας ρόλος είναι αυτόνομα να διδραματίσουμε με το ρόλο του ειρηνοποιού, που είναι απαραίτητο σε αυτόν τον κόσμο. Ελπίζω αυτή η πηξίδα, όπως την αποκαλούμε, ε, να μας φανεί χρήσιμη τώρα που θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτά τα χαρτογράφητα νερά στο επόμενο διάστημα και βασίζομαι πάνω σας για τη συνεργασία και με άλλα θεσμικά όργανα και την καλύτερη εξοποίηση των δυνατοτήτων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Τώρα, στην ημερησία διάταξη έχουμε την ε, δήλωση της ύπατης εκπροσώπου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Επομένως, θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Μογκερίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο λαός της ε, Βενεζουέλας έχει αντιμετωπίσει και εξοπλιστεί να αντιμετωπίζει μια δραματική κατάσταση. Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. 7 εκατομμύρια ε, πολίτε στη χώρα χρειάζονται βοήθεια. 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι υποσυτίζονται σύμφωνα ε, με το ΦΑΟ και το UNHCR. 4 εκατομμύρια Βενεζολάνοι ήδη έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τέσσερα τελευταία χρόνια και οι μελλοντικέ προβλέψει μα δείχνουν σε συνεχεί αυξήσει. Ο περιφερειακό αντίκτυπο κρίση είναι πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά και τη σταθερότητα τη περιοχή. Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση αυθαίρετα έχει συλλάβει πολλά μέλη τη Εθροσυνέλευση ε, και ήρε την βουλευτική του ασυλία η περίπτωση του ε, καπετάνιου Ραφαήλα Κώστα ε, αφού συνελήφθη από τις ε, αστυνομικέ δυνάμει, από τι δυνάμει ασφαλεία, είναι σοκαριστική. Καλούμε για μια εξάρτητη έρευνα που να οδηγήσει του ηθήνοντε στη δικαιοσύνη. Είδαμε όλη την έκθεση της ε, κυρίας Μπασελέ, της είπα Προσωπείται για τα ανθρωπίνα δικαιώματα που επιβεβαιώνει ότι οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισραήλ είναι σοβαρέ και συχνέ. Υποστηρίζουμε πλήρω και τα απορίσματα τη έκθεση και τι συστάσει τη έκθεση εξέδωσα σήμερα μία δήλωση εκ μέρους και των 28 κρατών μελών δηλώνοντας ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την ε, είπατε πρόσωπο του ΙΕ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις προσπαθίες της για να διασφαλίσει ότι προστατεύονται πλήρως τα δικαιώματα των Βενεζολάνων. Υπό το φως της έκθεσης είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εργασίες προς το να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα για όσους εμπλέκονται σε πραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε βασανιστήρια, το να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική και κοινωνική εκτακτή κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι επίγον. Τις τελευταίες εβδομάδες κάτι άρχισε να κινείται σε διπλωματικό επίπεδο. Οι συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση της Νορβηγίας ξεκίνησαν στα Βαρβάντος την περασμένη εβδομάδα και τώρα που μιλάμε υλοποιείται μία νέα συνάντηση. Ξέρουμε ότι ο δό προς τη δημοκρατική μετάβαση είναι σπαρμένη με εμπόδια. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά τις τελευταίε μήνες ή χρόνια μπορεί αυτό να είναι ένα πρώτο βήμα προ την ορθή κατεύθυνση προς μια ειρηνευτική και δημοκρατική μετάβαση με ελεύθερε και αξιόπιστε προεδρικές εκλογές. Είμαι ε, περήφανη για τον ρόλο κλειδί που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Όταν η βία φαινόταν ε, ότι ήταν το μόνο παιχνίδι και μάλιστα πολύ επικίνδυνο, όχι μόνο για τη Βενεζουέλα, αλλά και για την περιοχή και τον υπόλοιπο κόσμο, εμεί επεμέναμε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για την κρίση και ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα έπρεπε να είναι και ειρηνικό και δημοκρατικό. Γι' αυτό συστήσαμε την ε, ε, Διεθνή Ομάδα Επαφής με την ε, συμμετοχή τεσσάρων χωρών της Λατινικής Αμερικής και μια πέμπτη χώρα από την περιοχή ζήτησε να μπει την προηγουμένη εβδομάδα. Το Contact Group ποτέ δεν υποτίθεται ότι θα διαμεσολαβήσει στις συνομιλίες. Το ξέραμε αυτό από την αρχή γιατί μια τόσο πολύπλοκη διαμεσολάβηση δεν μπορεί να γίνει από μια ομάδα και επειδή ξέραμε πολύ καλά ότι οι συνθήκες για να ξεκινήσει η διαμεσολάβηση όταν αρχίσαμε συστήσαμε την Διεθνή Ομάδα Επαφή, δεν υπήρχαν καθόλου. Έτσι λοιπόν η ομάδα δεν δημιουργήθηκε για μια διαδικασία διαμεσολάβηση. Ε, πάντοτε ήμασταν σαφείς σε αυτό. Ο ρόλο του Contact Group ήταν να προσπαθήσει να συνεισφέρει στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ξεκινήσει μια διαμεσολάβηση που να έχει νόημα στο κατάλληλο πλαίσιο και με αξιόπιστο τρόπο. Και τονίζω, ε, αυτό έγινε όταν φαινόταν σχεδόν αναπόφευκτη κλιμάκωση. Τώρα, έχουμε κάποιους μήνες καλής δουλειάς και θέλω να ευχαριστήσω και τους Υπουργούς Εξωτερικών ε, των ε, χωρών της Ελληνικής Αμερικής αλλά και των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και τα μέλη της ομάδας που δουλεύουν μέρα νύχτα με πάρα πολλή αφοσίωση. Μετά λοιπόν από μήνες εργασιών ε, σήμερα μια δυνατότητα να οικοδομηθεί μια δημοκρατική και ελληνική λύση έχει ανοίξει. Ε, ο ρόλος ε, της ομάδας επαφής έχει αναγνωριστεί από όλα τα μέρη και εντός της χώρας και στην περιφέρεια αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι με όλους τους ε, διεθνείς συνομιλητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία ως την Κίνα, από το Βατικανό μέχρι την Κούβα, από την ομάδα της Λίμας μέχρι την Καρικόμη. Οι εκπρόσωποι της Contact Group συνάντησαν όλους τους ε, ε, πρωταγωνιστέ από τη Βενεζουέλα στο Καράκα. Ο Ερίκη Εγκλέσια ήταν στη Βενεζουέλα πριν λίγε μέρε και συνάντησε σε υψηλότερο επίπεδο όλους τους αρμοδίους, το Γουάν Γαϊδό, τον Νικολάς Μαδούρο, ε, τα Ηνωμένα Έθνη, τα κύρια πολιτικά κόμματα, αλλά και προσώπους της Καθολικής Εκκλησίας και της κοινωνίας των πολιτών. Η δουλειά αυτή ήταν ζωτική για να, ξεκινεί, να ανοίξει το χώρο για μια πολιτική λύση. Βέβαια δεν θεωρείται καθόλου δεδομένο ότι ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί για να πετύχουμε μια πολιτική λύση αλλά τουλάχιστον έχουμε σταματήσει την κλιμάκωση της στρατιωτικής βίας και έχουμε δώσει μια ευκαιρία στην πολιτική λύση. Γι' αυτό όλοι συμφωνήσαμε στην Κωνσταντίνα πριν λίγους μήνες στη συνάντηση του Contact Group να συνεχίσουμε τις εργασίες μας αλλά και να αντιδικοποιήσουμε την πολιτική μας δέσμευση και την απευθυνσή μα σε διάφορου διεθνεί ε, παράγοντε. Η διαδικασία που ξεκίνησε τώρα είναι πάρα πολύ εύθραστη. Όμω, ακριβώ γι' αυτό θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μα τώρα για να υποστηρίξουμε τι συνομιλίες στο Μπαρμπάιντο. για μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση πρέπει να έρθει από το εσωτερικό τη Βενεζουέλα. Ποτέ δεν μπορεί να επιβληθεί από το εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία με κάθε μέσο, όπω κάναμε του τελευταίου μήνε και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η χώρα χρειάζεται νέες προεδρικές εκλογές με μια ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία με ίσους κανόνες για όλους τους υποψηφίου. Επίσης, η χώρα χρειάζεται διάκριση των εξουσιών, ξεκινώντας από την αναγνώριση και το σεβασμό των προνομίων των ε, Εθνικών Συνελεύσεων και με συλλεία για όλα τα μέλη. Κάποια ουσιαστικά στοιχεία για μια αξιόπιστη διαδικασία έχουν αναδειθεί με σαφήνεια από τις συνομιλίες ε, και από τις εργασίες μας τους τελευταίους μήνες. Καταρχήν ε, ότι το ανώτατο δικαστήριο και άλλα όργανα πρέπει να εργάζονται για όλους τους πολίτες αμερόληπτα στη Βενεζουέλα και πρέπει να ε, υπάρχει μια νέα σύνθεση του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου. Δεύτερον, όλες οι υποψήφοι επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εκλογές με τα ίδια δικαιώματα και με, χωρίς να υπάρχουν αυθαίρετοι περιορισμοί. Τρίτον, ε, να επικοινωνηθεί το μητρό των ψηφοφόρων, να συμπεριλάβει και τους νέους ψηφοφόρους και τους κατοίκους εξωτερικού. Τέταρτον, ε, οι παρατηρητές ε, να παρακολουθούν όλη την εκλογική διαδικασία και όχι μόνο τις ημέρες των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Contact Group είναι έτοιμα να βοηθήσουν σε όλη την εκλογική διαδικασία αν ζητηθεί υποστήριξή μας από τα μέρη και να φτάσουμε στο στάδιο αυτό. Πιθανότατα αυτή είναι η πιο λεπτή στιγμή ε, σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική και δημοκρατική διαδικασία. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε όσο μπορούμε για να ενδυναμώσουμε αυτή την εύθραστη διαδικασία και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις προσδοκίες ε, του λαού της Βενεζουέλας. Πρέπει να διατηρήσουμε ένα βαθμό πίεση. Το καθεστώς της Βενεζουέλας πρέπει να κατανοήσει ότι το status quo δεν είναι επιλογή δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι καλό για τη χώρα, ούτε για τους πολίτες, ούτε για την περιοχή, ούτε για τον κόσμο. Σήμερα με τις δηλώσεις μας, όπως συμμετέχουν και τα 28 κράτη-μέλη, υπενθυμίσαμε ότι και παραθέτω, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα διευρύνει τα στοχευμένα μέτρα. Ταυτόχρονα ξεκαθαρίσαμε εκ νέου και παραθέτω ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να ανατραπούν ε, σε περίπτωση που γίνει σημαντική πρόοδος προς την αποκατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέσω του Contact Group και σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ για να εγγυηθούμε πλήρη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς, ε, ούτε ε, στι τοπικέ ΜΚΟ. Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση που ε, προωθήσαμε αυτού του μήνε και με του διορισμούς του, και με το διορισμό του συντονιστή από τον ΟΗΕ. Από την έναρξη της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήμασταν ε, ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα και εντός ε, της χώρας αλλά και στις όμορες χώρες. Συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο κάθε περιφερειακή και διεθνή πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί η κρίση των προσφύγων ξεκινώντας με τη διαδικασία του Κίτο. Και αυτό δεν θα αλλάξει καθώς εργαζόμαστε επί του πολιτικού θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ ενεργοί στην ανθρωπιστική στήριξη. Όμως πέρα της ανθρωπιστικής βοήθειας νομίζω ότι έχουμε και την ευθύνη να συνεχίζουμε ε, να παρακολουθούμε ε, τις εργασίες για να υπάρξει μια διέξοδος από την κρίξη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρανζέλ, εκ μέρους του ΕΛΚ, για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία, είπατε εκπρόσωπα. Εγώ θεωρώ θεμελιώδες ότι την πρώτη στιγμή αυτής της θητείας όταν ξεκινούν οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουμε μια σαφή θέση σε σχέση με την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Είναι θεμελιώδες αυτό να είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλέπουμε βασανιστήρια, δολοφονίες, πολιτικές διώξεις. Ε, που λαμβάνουν χώρα κατά των ε, αντιπολιτευόμενων. Επίσης υπάρχουν ε, επιθέσεις κατά της Εθνοσυνέλευση, κατά της πολιτικής ελευθερίας έκφρασης και ταυτόχρονα να αναγνωριστεί η Εθνοσυνέλευση και ο Χουάν Γουαϊδό ως συνόμιμη εκπρόσωποι του λαού της Βενεζουέλας. Λεχθέντων αυτών είναι πολύ σημαντικό επίσης να, προ... να πείσουμε τις αρχές ε, να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε την μεταναστευτική κρίση στο Εκοδόρ, στην Κολονδία, στο Περού, ακόμα και στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, όπου κάθε φορά έχουμε πολύ περισσότερους πολίτες από τη Βενεζουέλα. Έχουμε τη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση στην Αμερικανική Ήπειρο και είναι σημαντικό να ευστήσουμε την προσοχή για ε, την απαράδεκτη ε, παρέμβαση της Κούβας και της Ρωσίας. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η διαδικασία του διαλόγου ε, όπου διαμεσολαβεί η Νορβηγία και θα πρέπει να έχουμε στόχο την υλοποίηση διαφανών δημοκρατικών ελεύθερων εκλογών όπου θα τοποθετηθεί κυρίαρχα ο λαός της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Λόπες, για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την είπατε εκπρόσωπη. Εμεί συμφωνούμε με την ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη είπατε εκπρόσωπη για την Βενεζουέλα. Όμω θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα να τονίσουμε την αλληλεγγύη μας ε, με το λαό τη Βενεζουέλας και να πούμε ότι η μόνη διέξοδος είναι η ειρηνική πολιτική και αποδιαπραγμάτευση που θα καταλήξει σε ελεύθερες και δίκαιε εκλογές με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολιτικούς πρωταγωνιστές και με παρατηρητές από τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να διεκδικήσουμε να υπάρχουν τώρα θετικές ε, προσδοκίες που στα με τη διαμεσολάβηση της Νορβηγίας υλοποιούνται οι διαπραγματεύσεις αυτές. Και επίσης είναι η στιγμή να ε, ρίξουμε το φως για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Στα δεινά που υποφέρει ο λαός και στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Μπασελέτ. Έχουμε εξοδικαστικέ εκτελέσει, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανιστήρια με τιμωρησία και πρέπει να απαντηθούν αυτό. Και επίση έχουμε παραβίαση σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Για όλα αυτά, εμεί σήμερα θέλουμε να ε, παρουσιάσουμε τη μοναδική διέξοδο και ταυτόχρονα ε, να παρουσιάσουμε τα δεινά που βιώνει ο λαός της Βενεζουέλας. Και να πούμε τώρα ότι μόνο χάρη στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκ μέρους ομάδας Renew Europe η Αντιπρόεδρος κυρία Σαράτσοβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ είπατε, είπατε εκπρόσωπε, αύριο είναι η μέρα της ε, παγκόσμιας, ε, της διεθνούς ποινική δικαιοσύνης. Δεν ενεχόμαστε στη Βενεζουέλα να παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μια πιο κάθετη θέση απέναντι στη δικτατορία και να διευρύνει τις επιλεκτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις και στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία. Λένε ότι ο Μαδούρο είναι διτεθειμένος να διαπραγματευτεί. Όμως εγώ αναρωτιέμαι πώς ε, κάποιος ε, μπορεί αφενός να διαπραγματεύεται και αφετέρου την ίδια στιγμή να φυλακίζει, να βασανίζει και να δολοφονεί τους ε, αντιπολιτευόμενους στο καθεστώς, πώς είναι δυνατόν να λέει ότι θέλει διάλογο και ταυτόχρονα να διώκει αυτούς ε, με τους οποίους υποτίθεται θέλει να διαπραγματευτεί. Ας μην απατώμαστε το Μαδούρο, συνεχίζει ε, πάντοτε να κάνει τα ίδια τρίκ και θέλει να κερδίσει χρόνο. Ε, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να διασφαλίσουμε ότι ο Μαδούρο τελικά θα δεσμευτεί σοβαρά στην υλοποίηση του διαλόγου και ότι η κρίση θα επιληθεί ειρηνικά. Ευχαριστώ.